και θα περάσουμε τώρα στην εκλογή των αντιπρόεδρων. Όσον αφορά την εκλογή των αντιπρόεδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνω να ορίσουμε μία προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιωτήτων για τις μία το μεσημέρι. Μία το μεσημέρι είναι η προθεσμία. Ελπι... Παρακαλώ να δώσετε τις υποψηφιώσεις αυτό στο R00111 στα χέρια του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέου. Είναι το γραφείο της ε, Προεδρίας το κτίριο Λουίς Βάις. Επί διαδικασία δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Διακόπτω λοιπόν εδώ τη συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε στις 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.